που υπέγραψε τους στόχους της χιλιτίας μέχρι που μετά άρχισε να το σκέφτεται στο δρόμο της επιστροφής στο αεροπλάνο. Και μετά άρχισε να σκέφτεται ότι α, δεν βαριέσαι, άλλη μια δήλωση. Και μετά συνέχισε λέγοντας λέγοντας ότι δεν μπορούσα να κάνω μεγαλύτερο λάθος και έδωσε συγκεκριμένα παραδείγματα για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί. Κάποιοι στόχοι έχουν επιτευχθεί, κάποιοι τους έχουμε υπερβεί. Υπάρχουν άλλοι όμως που δεν έχουν επιτευχθεί. Πάντως εν γέννη το να έχουμε θεσπίσει ένα μικρό αριθμό στόχων σήμανε σημαντική πρόοδο και υπάρχει ακόμα χρόνος για να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο. Το σημαντικό θέμα είναι ότι το επόμενο, η επόμενη φάση θα πρέπει όντω να μα οδηγήσει στην την βιώσιμη ανάπτυξη. Όμως, για να γίνει αυτό, πρέπει να ε, μας, ε, να μας ε, υποστηρίζουν και οι λαοί μα και ίσω αυτό να είναι ενδιαφέρον για του συναδέλφου από τα κοινοβούλια που μα επισκέπτονται τώρα. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι είμαστε σε αυτή την περιοχή η ύφεση λιτότητα, διαρκώ περικόπτονται οι μισθοί, οι συντάξει μειώνονται οι υπηρεσίε, αυξάνονται οι φόρες σε όλες μας τις χώρες για να βάλουμε μια τάξη και να ελέγξουμε τη δημόσια οικονομία μα. Και από αυτέ τι ε, περιστάσεις υπάρχει κόσμος που βλέπει τον, στο, τον, τον ε, προϋπολογισμό, τον αναπτυξιακό, καθώς και τις ε, ε, προσπάθειες που κάνουμε για να βοηθήσουμε τον αναπτυσσόμενο κόσμο ως κάτι το οποίο που δεν μπορούμε τελικά να κάνουμε στην πράξη. Όμως ο κόσμος τελικά είναι πολύ γενναιόδρος και αν μιλήσουμε για τις επιτυχίες μας θα ανανεωθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου, θα συνεχίσει να θέλει να βοηθήσει. Όταν ε, ας πούμε πάω σε κάποια λέσχη νέο να μιλήσω ή ε, οι επιχειρηματίες βρίσκουν τον τρόπο να εισάγουν περισσότερη εργασία για την Επιτροπή Ανάπτυξης ή για την αντιπροσωπεία. Εγώ πάντοτε λέω δύο πράγματα. Ε, ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό ότι καθημερινά 23.000 γυναίκες και παιδιά πεθαίνουν στον αναπτυσσόμενο κόσμο αλλά απ' την άλλη είναι εντυπωσιακό και ενθαρρυντικό το ότι οι άλλες 23.000 δεν πεθαίνουν πια. Ας κάνουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε για να μειωθεί ακόμη περισσότερο κόσμο. και βλέπεις πάντα κόσμο στο ακροτήριο που θέλει, βλέπει με ενθουσιασμό όλα αυτά. Αν διαρκώς ε, ε γκρινιάζουμε και θρυνούμε και απελπιζόμαστε, ε, τότε και ο κόσμος απελπίζεται. Τελικά λοιπόν αποκόμισα μια αίσθηση από αυτήν την διάσκεψη κορυφής για τους στόχους της χιλιετίας ότι έχουν γίνει πολλά, αλλά ότι μπορούμε και να βασιστούμε σε αυτά που έχουν ήδη γίνει για να επιτύχουμε και άλλα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι δεν το κάνουμε αυτό μόνο για ανθρωπιστικούς λόγους, αλλά και για εγωιστικούς λόγους. Γιατί όπως εμείς στην Ευρώπη προσπαθούμε να δικοδομήσουμε την ειρήνη και τη σταθερότητα βοηθώντας ένα τον άλλον, πρέπει να κάνουμε το ίδιο και στον υπόλοιπο κόσμο που αλλάζει διαρκώς και θέλουμε να έχουμε καλές σχέσεις και επαφές. Υπάρχουν δηλαδή και εγωιστικοί και αγνοί λόγοι για τους οποίους προσπαθούμε να κάνουμε όλα αυτά. Ε, έγινε πολλής λόγος για διαφάνεια και η διαφάνεια είναι ένα σημαντικό κομμάτι των προσπαθειών της ε, κοινότητας της αναπτυξιακής. Πρέπει να μετακινηθούμε νομίζω από την, την διαφάνεια σε σαφείς μηχανισμούς λογοδοσίας, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνονται πράγματα και ότι όταν θα θεσπίζονται στόχοι θα υπάρχει ένας μηχανισμός αναφοράς. Ε, να δούμε δηλαδή αν όντως επετεύθηκαν οι στόχοι που είχαμε θέσει και αν όχι γιατί. Ε, πολλά βέβαια πρέπει ακόμα να γίνουν, αλλά έχουμε την αίσθηση πως η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι στιγμής άξιζε τον κόπο και θα πρέπει να εξακολουθήσουμε να παίζουμε ισχυρό και επικοδομητικό ρόλο στις επερχόμενες διαπραγματεύσεις. Σας ευχαριστώ. Πρόεδρος, σας ευχαριστώ πολύ και εγώ που μας ενημέρωσες για αυτή την εμπειρία και τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Κόρτες Κάστρα. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Συμμερίζομαι με τον κύριο Μίτσελ φυσικά ότι μια αντιπροσωπεία σημαντική και που πιθανόν και στην δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή έφερε πιο κοντά το πώς έχει ανάπτυξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας που θα είναι πάντα σημαντικό θέμα για την Επιτροπή μας να έχουμε τέτοιου είδους επαφές, διμερείς επαφές ε, όπως ε, ε, σε αυτό το πλαίσιο. Χωρίς αμφιβολία βρισκόμαστε σε μια στιγμή που πρέπει όχι να μειώσουμε τις προσπάθειες για τους στόχους αλλά πρέπει να καταλήξουμε στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Το έγγραφο αυτό είναι ένα αποδεκτό έγγραφο, αλλά μπορεί να δημιουργήσει όμως κάποιες ανησυχίες ακόμα. Λοιπόν πρώτον, για τους επόμενους 15 μήνες αφήνουμε στα χέρια κυβερνήσεων αποκλειστικά την τελική ανάπτυξη του τελικού εγγράφου για την ανάπτυξη των στόχων της χιλιετίας. Και αυτό για τη χώρα μου, για μένα, για το τι συνέβη με την δική μας κυβέρνηση και την περικοπή των κονδυλίων για την ανάπτυξη, δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε την προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις διαπραγματεύσεις που θα γίνουν τους επόμενους μήνες. Και γιατί το λέγω αυτό, διότι σε αυτή την αντιπροσωπεία στη Νέα Υόρκη είχαμε μια θέση στεναρή και συνενετική για την ανάπτυξη, συνεργασία για την ανάπτυξη και όπως είπε, ακούστηκε από πλευράς Προέδρου, βασιζόμαστε σε τέσσερις αρχές. Την παγκοσμιότητα, την διαφάνεια, τη συμμετοχή των ε, πολιτών, την αποτελεσματικότητα. Προσέξτε όμως, η Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να επιτρέψει σε καμιά περίπτωση αυτό να μετατραπεί σε ένα ευχολόγιο, σε ένα κατάλογο ευχών όπως κάνουμε τα Χριστούγεννα. Το αντίθετο πρέπει να επικεντρώσουμε κάθε προσπάθεια να είναι συγκεκριμένες μετρητές, μετρήσιμες αυτές οι προσπάθειες για αυτά τα μέτρα και ή δυνατόν ευχόμαστε να είναι δεσμευτικού χαρακτήρα για τα επόμενα χρόνια. Εγώ ειλικρινά και σε σχέση με τις δικές σας χώρες, εγώ δεν πρέπει να μιλήσω μόνο για τη χώρα μου, αλλά και για κάτι το οποίο με ενοχλεί βαθιά. Είδαμε αυτά τα χρόνια, κυρίως αυτά τα τελευταία χρόνια πρόσφατα, πως χωρίς να υπάρχει κανένα εμπόδιο αυτή η κοινωνία <clears throat> για την υπέρβαση των, ε, των ε, υπηρεσιών που έπρεπε να ληφθούν υπόψη κάναμε ό,τι έπρεπε και όμως βλέπουμε να υπάρχουν ακόμα πολλές επιφυλάξεις πολλές επιφυλάξεις και ενδιασμοί για τη συνένεση και την δημιουργία ενός προγράμματος ε, με στόχους μετρήσιμους, συγκεκριμένους και ή δυνατόν και δεσμευτικού χαρακτήρα ακόμα κιόλα. Και ολοκληρώνω η ανισότητα όχι μόνο στον παγκόσμιο, στον κόσμο σημειώνεται αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Η φτώχεια δεν είναι μόνο κάτι που σημειώνεται σε άλλες χώρες παγκόσμια αλλά και εδώ στην Ευρώπη. Και ως προς αυτό εμείς ως Ευρωβουλή πρέπει με μεγαλύτερη υπευθυνότητα να αγωνιστούμε για την καταπολέμηση της φτώχειας αλλά και εδώ στο ίδιο το Ευρωκοινοβούλιο για την καταπολέμηση της φτώχειας στην Ευρώπη και μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη περισσότερο ακόμα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Θα λάβει τον λόγο ο κύριος Τέιλορ παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο ομιλητής. I would like to say thank you very much. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη γραμματεία που διοργάνωσε το ταξίδι και για το, στον κύριο και για την έκθεσή του. Θα ήθελα να κάνω μόνο ένα μικρό σχόλιο. Ξέρω ότι έχουμε περιορισμούς όσον αφορά την επιλογή των μελών που θέλουν να πάνε στις διάφορες αντιπροσωπείες, αλλά είχαμε μια αντιπροσωπεία, ε, μια μελή και, και όλοι πήγαν. Πράγμα το οποίο μας έκανε να πάμε εκεί και να ακούσουμε τα σχέδια για αύξηση της χειραφέτησης των γυναικών και ισότητα των φύλων, αλλά τελικά ε, χωρίς να έχουμε τη δυνατότητα να αισθανθούμε την ισορροπία των φύλων ε, στην οδηγία μας την ίδια την αντιπροσωπεία. Γι' αυτό και ήμασταν λίγο σε δύσκολη θέση κάποιες φορές. Ίσως θα έπρεπε να υπάρχει κάποια ενθάρρυνση από πλευρά των ομάδων, ώστε να υπάρχει ισορροπία ε, φύλων στις αντιπροσωπείες. Επανέρχομαι στην ίδια την διάσκεψη και ως νέο μέλος αυτής της Επιτροπής δεν μπορούσα παρά να εντυπωσιαστώ από τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν όλες οι συζητήσεις. Οι υφιστάμενοι στόχοι της χιλιτίας φαίνεται ότι λειτουργήσαν ως όθηση ε, για τις κυβερνήσεις και για τις ΜΚΟ. Ε, οι δε κυβερνήσεις είναι υπόλογες στο γεγονός ότι υπάρχουν στόχοι και ότι πρέπει να επιτευθούν. Οι στόχοι της χιλιτίας λοιπόν ως έχουν άξιζαν τον κόπο. Φυσικά υπήρξαν ε, κάποια στοιχεία που δεν ήταν ακριβώς όπως ε, θα επιθυμούσαμε ή θα είχαμε ελπίσει, αλλά θα ήταν ε, ιδανικό να καταλάβουμε και να μάθουμε για τη θέσπιση των στόχων του 2015 και ιδιαίτερα η ανάπτυξη αυτών των στόχων θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς γιατί έχω διάφορα σχόλια ότι δηλαδή τη διαδικασία δεν θα πρέπει να την ιδιοποιούνται μόνο οι πλούσιες χώρες ε, και να ε, υπαγορεύουν στις στοχές χώρες το τι είδους ανάπτυξη χρειάζονται. Αυτό ήταν αρκετά ισχυρό μήνυμα σε αυτή την ιδιαίτερη εκδήλωση. Οι στόχοι της χιλιετίας που επετέφθησαν ή εν μέρη επετέφθησαν, δηλαδή η μείωση της παγκόσμιας στόχιας, η εκπαίδευση, έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια και μεγάλα βήματα στην υγεία για την ελονοσία και τη μείωση του AIDS κάποιες ε, από τους λιγότερο καλούς ε, στόχους ήταν ε, η θνησιμότητα η παιδική, βιωσιμότητα και οι παγκόσμιες εταιρικές σχέσεις για την ανάπτυξη. Τώρα, το έγγραφο των πορισμάτων αυτής της ειδική ε, διάσκεψης δείχνει ότι χρειάζεται μία επιπλέον και τελική προσπάθεια ώστε παγκόσμια να βελτιώσουμε την απόδοσή μας για την επίτευξη αυτών των στόχων και όλος ιδιαίτερος να πούμε στη, να δούμε μάλλον στην ημερήσια διάταξη για μετά το 2015 εγώ βρήκα πως ήταν χρήσιμο να έχουμε τρεις τρία, τρεις ειδικές επιτροπές πάνελ, ένα εκ των οποίων ήταν η ανάπτυξη βιώσιμων ρυθμίσεων για χρηματοδότηση, ώστε να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους μετά το 2015. Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες. Η ιδέα είναι να συνδυαστεί η κρίση της στόχης με, την βιώσιμη, με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το 2020. Δεν μπορεί κανείς να αφιβάλλει πως τα δύο αυτά είναι αλληλένδετα. Κανένα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς το άλλο. Επίσης ακούσαμε την χειραφέτηση και την ισότητα των φίλων. Πρέπει να πούμε ωστόσο ότι δεν αναφέρθηκε καμία, κανενός είδους συμφωνία όσον αφορά το θέμα των ομοφιλοφίλων. Οι πόρτες ήταν αυστηρά κλειστές όταν προσπαθήσαμε να θίξουμε θέματα ε, που αφορούν τους ομοφυλόφιλους. Σε πάση περιπτώσει πρέπει να προχωρήσουμε με αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Μιλήσαμε λοιπόν για την προώθηση των γυναικών στην ε, γεωρική παραγωγή, ιδιαίτερα μέσω του προγράμματος ε, των, παγκοσμίων προγραμμάτων για την, τα τρόφιμα υπάρχει μια πρόκληση που μας υπέβαλε ο Μπαν Κιμούν ε, για μηδενική πείνα, δηλαδή ανάπτυξη μικρής κλίμακας ε, τοπικών ε, δικτύων παραγωγής τροφίμων. Αυτά είχα να πω, νομίζω. Και να πω επίσης ότι έχω την εντύπωση, όπως και ο Γκέι, πως υπάρχει αποφασιστικότητα να μάθουμε από τα λάθη της διαδικασίας της τωρινής, της τρέχουσας για τους στόχους χιλιετίας και να δουλέψουμε με πιο συνολικό, διάφανο ε, τρόπο με έλεγχο και παρακολούθηση και να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε παγκόσμια ένα οικονομικό κλίμα και και λόγος για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Εγώ, Εγώ προσωπικά δεν είμαι πολύ πεπισμένος γι' αυτό. Πάντως έγινε λόγος για την ε, ένταξη καινοτόμων οικονομικών ε, καινοτόμου μάλλον οικονομική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτό. Θα, δω, θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει και θα κάνω σίγουρα ό,τι μπορώ για να προωθήσω τους στόχους όπως θα προκύπτουν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα σε σχέση με αυτό να αναφέρω ότι πρώτον θεώρησα ότι αυτή η αποστολή ήταν πάρα πολύ διδακτική και ενδιαφέρουσα. Πραγματικά επί τόπου μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Πολύ συχνά κατανοεί καλής, κανείς καλύτερα επιτόπου τα θέματα, έρχεται σε επαφή με τους άμεσα εμπλεκόμενους, κατανοεί έτσι λοιπόν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι σημαντικό αυτό για να καταλάβει κανείς τους λόγους και την αιτιολογία που βρίσκονται πίσω από μια συγκεκριμένη κατάσταση και ένα πρόβλημα. Μπορώ να πω ότι η συνεργασία στην αντιπροσωπεία μας ήταν πραγματικά πολύ επικοδομητική. Ευχαριστώ ιδιαίτερα επίσης και την γραμματεία πρέπει να πω για τη διοργάνωση των πραγμάτων. Οργανωτικά είχε προπαρασκευαστεί η αποστολή εξαιρετικά. Αυτά που ήθελα να πω τα προανέφερε ο συνάδελφος Τέιλορ. Εννέα μέλη της αντιπροσωπείας μας, εννέα άνδρες είμαστε από την αντιπροσωπεία μας. Δίνεται όμως μια πολύ αρνητική εικόνα με αυτή τη σύνθεση ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το γνώριζα θα είχα εγώ αποσύρει τη δική μου υποψηφιότητα και θα είχα προτείνει μια συνάδελφος Ευρωβουλευτή να συμμετείχε σε αυτή την αποστολή. Θα είχαμε τουλάχιστον μία συνάδελφο σε αυτή την αποστολή, ίσως από την Επιτροπή Δικαιωμάτων των γυναικών και ισότητα των φίλων θα μπορούσε να γίνει αυτό. Μελλοντικά θα πρέπει να μας προβληματίσει αυτό, να δούμε πώς θα μπορέσουμε σε τέτοιες αντιπροσωπείε να συμμετέχουν και γυναίκες και να μην συμμετέχουν μόνο αποκλειστικά άνδρες. Πάει αυτό για αυτό το σημείο, επόμενο σημείο για την έκθεση. Στην έκθεση εμπεριέχονται πολλά καλά πράγματα, όμως καμιά φορά αυτή η έκθεση περιγράφει μια συνενετική κατάσταση των πραγμάτων και είναι κάπω προβληματικό αυτό, διότι δεν είναι πάντα δεδομένο ότι είμαστε, έχουμε συνένεση επί κάποιων θεμάτων πάντα. Υπάρχουν κάποια θέματα για τα οποία δεν συνενούμε όλοι απόλυτα. Δεν έχω καμιά αντίρρηση να αναφέρετε κάτι τέτοιο, αλλά πρέπει να αποσαφηνίστε ότι έχουμε και διαφορετικές απόψεις επί κάποιων θεμάτων, όπως για τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, για παράδειγμα, ή σε σχέση με τα αποτελέσματα όσον αφορά του ε, περιβαλλοντικού στόχου. Μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από όσα αναφέρθηκαν από τον κύριο Μίτσελ κτλ. ότι τα θετικά πρέπει να θέσουμε στο επίκεντρο και στο προσκήνιο. Όμως από την άλλη πλευρά και τα αρνητικά σημεία θα πρέπει να μπορούν να αναφέρουν οι στόχοι εκείνοι οι οποίοι δεν επετέφθησαν μέχρι τούδε. Η ισότητα για παράδειγμα. Μέχρι σήμερα δεν καταφέραμε πολλά πράγματα. Τίποτα δεν καταφέραμε για την ισότητα. Δεν βελτιώθηκε η θέση των γυναικών όσον αφορά τα ίσα δικαιώματα όσο σε σχέση με πριν από 10 χρόνια όταν ε, προχωρήσαμε στους στόχους της χιλιετίας ε, τότε. Και θα ήθελα να πω ότι κάπως πρέπει να πω με εκπλήσει το γεγονός ότι στην έκθεση αυτή κάποια πράγματα έχουν παραμείνει εκτός, απουσιάζουν. Προσπάθησα κάποια σημεία να τα αναφέρω. Έγινε αυτή η προσπάθεια. Δεν μιλήσαμε μόνο για την αναπαραγωγική υγεία, τα δικαιώματα ε, τα, και, τα θέματα τα, τα σεξουαλικά και τις, ε, τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Κάναμε μεγάλο λόγο, πολύ λόγο για αυτά τα θέματα. Αυτό όμως αποτελεί τη διαφορά. Δεν είναι το θέμα να γίνεται μόνο λόγος αλλά το θέμα είναι να δούμε ότι σε κάθε συνεδρίαση, σε κάθε συνάντηση ε, για τα δικαιώματα και για την ε, δυνατότητα διαμόρφωσης των δικαιωμάτων αυτών θα πρέπει να γίνεται λόγος και αυτό πρέπει να αναφέρεται. Καλό θα ήταν λοιπόν αν θα μπορούσαμε εδώ να αναφέρουμε αυτό το οποίο όλοι οι ευρωβουλευτές ανέφεραν και όχι αυτό το οποίο μόνο κάποιοι ανέφεραν και τοποθετήθηκαν επί κάποιων συγκεκριμένων θεμάτων γιατί διαφορετικά δημιουργείται εντύπωση ότι όλοι συμφωνούν διαφωνούν επί μερικών απόψεων. Επ' αυτού ασκώ επικρίσεις. Αν αυτό γίνεται τότε θα πρέπει να φαίνονται όλα τα θέματα τα οποία εθίγησαν και καλύφθηκαν από τους ευρωβουλευτές. Διότι πάρα πολλά θέματα αναφέρθηκαν και καλύφθηκαν και αυτό δεν είναι μια πολιτική έκθεση αυτό που έχουμε μπροστά μας. Πρέπει να είναι μια περιγραφή κατάστασης, περιγραφή δεδομένων. Και τώρα για το έγγραφο, το outcome document, το ε, ε, έγγραφο των αποτελεσμάτων και θέσεων. Ε, είναι πολύ σύντομο, υπερβολικά σύντομο. Υπάρχουν πολλά περιθώρια να μπορέσουν να συζητηθούν κάποια πράγματα και να εμβαθυνθούν κάποια πράγματα. Όμως έχουμε και θετικά πράγματα σε αυτό το τελικό έγγραφο. Και είναι καλό να μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι και κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα στόχοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν. Αυτό είναι ε, καλό. Δεν μπορούμε να κάνουμε λόγο για κοινωνικούς στόχους αν ταυτόχρονα δεν λαμβάνουμε υπόψη και τους οικολογικούς στόχους που πρέπει να είναι σεβαστοί. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα. Τέσσερα παραδείγματα θα ήθελα να αναφέρω στο θέμα των ίσων δικαιωμάτων. Δύο είναι θετικά, δύο είναι αρνητικά. Καλό είναι ότι το τελικό έγγραφο αναφέρει ότι η συνολική διαδικασία των στόχων ανάπτυξης της χιλιετίας ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη ε, και το, τη διάσταση ε, του φύλου και ότι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων είναι προϋπόθεση, αναγκαίος όρος και προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος με το γεγονός ότι το σύνολο θέμα, συνολικό θέμα των σεξουαλικών και αναπαραγωγικών δικαιωμάτων δεν αναφέρεται. Είναι σημαντικό εκεί. Σπουδαία αυτή η απουσία. Έχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Οι γυναίκες έχουν δικαίωμα να αποφασίζουν τι θα γίνεται με το σώμα τους, με τα σώματά τους. Και δεν ε, είναι δυνατόν να αναφέρετε ότι αποτελεί ένα ξεχωριστό ε, μόνο στόχο. Θα ήθελα αυτό να εμπεριέχεται εδώ, όχι μόνο να το αναφέρουμε. Θα ήθελα να υπάρχει δυνατότητα στο μέλλον να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτά και να εξειδικεύσουμε περισσότερο αυτά. Ξέρω ότι οι διαπραγματεύσει είναι δυσχερεί όταν ε, συμπεριλαμβάνονται τόσε πολλέ χώρε αυτέ. αυτά θέλω να πω ήταν θετικό να είμαστε επιτόπου, διότι μαθαίνει κανείς με αυτόν τον τρόπο επιτόπου περισσότερα και μαθαίνει και τις απόψεις των άλλων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μαρτίνες παρακαλώ, στη συνέχεια έχει τον λόγο. Θα σε ευχαριστώ πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι θέλω να επικεντρωθώ μόνο αποκλειστικά σε ένα θέμα. Όμως αυτό που είπε μόλις ο κύριος Γκούσταυσον, πρέπει να πω εντάξει συμφωνώ με τον κύριο Γκούσταυσον στις σκέψεις που εκφράζει. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι εγώ πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι ένα πολιτικό έγγραφο και δεν είναι τα πρακτικά αυτών που είπε κάθε ένας σε κάθε συνεδρίαση που είχαμε. Διότι Πρώτον, θα ήταν εκτενέστατο έγγραφο αν γινόταν κάτι τέτοιο. Δεύτερον, πρέπει να αναζητήσουμε εκείνα τα σημεία όπου υπήρξε συμφωνία και σημειώθηκε πρόοδος επ' Τώρα, εδώ θα ήθελα να πω το εξή. Ένα πράγμα έμαθα και ο κύριος Γκέι Μίτσελ το ανέφερε πιο πριν. Αν θέλω το πω με μεγαλύτερη ευκρίνεια, με μεγαλύτερη σαφήνεια, έμαθα ένα μάθημα σημαντικό σε αυτό το θέμα, που είναι ένα σημαντικό μάθημα. μάθημα. Και επίσης με εμπνέει, γι' αυτό αυτό που είπε η Πρωθυπουργό στην Νορβηγία τότε παλαιότερα. Πιστεύω λοιπόν ότι όλοι μας βρεθήκαμε σε μια δυναμική των πραγμάτων εσφαλμένη και επικίνδυνη επί μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτό διαρκώς ε, μας οδηγούσε στο να λέμε είναι μισογεμάτο ή μισοάδιο το ποτήρι και ακόμα περισσότερες φορές να λέμε και κάτι χειρότερο από μισοάδιο. Δηλαδή είχαμε πληροφορίες ακριβείς και σαφείς στη Νέα Υόρκη για το ότι σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος στο θέμα των διαφορετικών στόχων της ανάπτυξης, για την ε, ανάπτυξη της χιλιετίας. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και για μια ολόκληρη σειρά ετών, και ασκώ επίκριση σε αυτό, όλοι μας, οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις πρώτα απ' όλα, είμαστε οι υπεύθυνοι για τα πολιτικά θέματα σε αυτό το θέμα από πλευρά μα, αξιολογούσαμε με πολλέ επικρίσει και πολύ αρνητικό τρόπο το ότι δεν σημειωνόταν πρόοδο, πρόοδος, αυτό δεν θα οδηγούσε πουθενά, δεν πηγαίναμε, δεν σημειώναμε πρόοδο, έγιναν πολύ λίγα και δεν έγιναν αρκετά. Αυτό είναι μια λανθασμένη στρατηγική και επικίνδυνη στρατηγική και είναι μια στρατηγική που απόλυτα διευρύνθηκε και πολλαπλασιάστηκε από τα μέσα του τύπου και της ενημέρωσης που συνεισέφεραν στο να υποβιβαστεί αυτό το οποίο κάναμε και είχαμε και την έκπληξη εμείς οι ίδιοι επιτόπου να δούμε με αριθμιστικά στοιχεία, με αποδείξεις και στοιχεία τα οποία δεν χωρούν αμφισβήτηση ότι πραγματικά το ποτήρι ήταν πάνω από γεμάτο, Εντάξει, με φυσικά διαφορές μεταξύ χωρών μεταξύ τους και φυσικά με μεγάλες διαφορές όσον αφορά κάποιους από τους στόχους σε σχέση με άλλους από τους στόχους της χιλιετίας. Όμως φυσικά ένα από τα πράγματα που είδαμε είναι και δεσμευθήκαμε και εγώ το είπα αυτό, δεν θα ξαναπώ ποτέ, δεν θα ξαναπούμε ότι είναι άδειο ή αδειο. Όχι μισοάδιο, λέγαμε ότι ήταν άδειο το ποτήρι, όχι καν άδειο. Και πολλές από τις οργανώσεις μας, τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις, και με καλές προθέσεις συνεισέφεραν πολλές φορές στη διαβίβαση ενός μηνύματος ότι δεν γινόταν τίποτα, δεν καταφέρναμε τίποτα. Και έτσι λοιπόν ε, βλέπαμε και είδαμε ότι έγιναν αρκετά. Όχι επαρκή, δεν επαρκούν, αλλά έγιναν αρκετά πράγματα δεν πεθαίνουν τόσα παιδιά όσα παλιότερα. 15.000 λιγότερα ημερήσια. Και αυτό μας κάνει περισσότερο να καταβάλουμε προσπάθειες. Να μην ξεχνάμε ότι τα 15.000 όμως ζουν, ενώ δεν ζούσαν, δεν θα επιζούσαν στο παρελθόν. Αυτό είναι ένα μάθημα το οποίο πρέπει να συναγάγουμε, να μάθουμε από αυτό και να το προαγάγουμε. Και να δούμε ένα από τα στοιχεία σε σχέση με τις ε, αρνητικότερες επικρίσεις είναι σε σχέση με το έγγραφο που εγκρίθηκε στη συνδυασία διάσκεψη όπου εμείς οι ίδιοι συμμετείχαμε και αυτό το έγγραφο είναι πραγματικά παράδεκτο, λέγανε. Αυτό όμω το έγγραφο πρέπει να το αξιολογήσουμε σαν ένα έγγραφο το οποίο προσυπογράφουν 189 χώρε. Και 189 χώρε δεν μπορούν να συντάξουν το ίδιο έγγραφο που ο κύριο Γκούσταφ ή ο ίδιο εγώ θα θέλαμε να είχαμε ή να συντασσόταν. Είναι όμω αρνητικό να λέει κανεί ότι είναι απαράδεκτο αυτό το έγγραφο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τίποτα. Είναι ένα καλό έγγραφο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ω βάση για να σημειώσουμε περισσότερη πρόοδο με όλες τις ελλείψεις, ε, τα ελαττώματα. Αυτό είναι το μάθημα που έμαθα κυρία Πρόεδρε και αυτό θα ήθελα εγώ να μπορέσουμε να το συναγάγουμε ως μάθημα όλοι μας για να μην διαβιβάζουμε και περνάμε το μήνυμα στην κοινωνία διαρκώς ένα μήνυμα ότι αυτά που κάνουμε και δαπανούμε δεν συνεισφέρουν με κανένα τρόπο να σημειωθεί πρόοδος όπως θα ήταν αναγκαίο να συνέβαινε. Σε σχέση για τις κυβερνήσεις μας για παράδειγμα με την κυβέρνηση της ε, Ισπανίας λένε εντάξει αν αυτό δεν βοηθάει προχωρήσουμε, ε, τότε α υπάρξουν περικοπές. Δεν θα είναι σημαντικό αν γίνουν και περικοπές σε κάτι που δεν βοηθάει. Λοιπόν, να μην περνάμε ένα τέτοιο μήνυμα. Πολλά φυσικά απομένουν να γίνουν και πρέπει να γίνουν, αλλά αυτό ήταν μια αποκάλυψη για μέσα. Να, το, το μήνυμα το οποίο περνάμε δηλαδή ότι δεν ωφελούν όλα αυτά τίποτα ότι οι στόχοι της χιλιετίας για την ανάπτυξη ήταν μια παταγώδης αποτυχία δεν ήταν παταγώδης αποτυχία ήταν μια πολύ αποδεκτή επιτυχία ευχαριστώ ο κύριος Νιούτον Ντάν. Παρακαλώ, παρακαλώ, αν θα μπορούσατε να σε συντομότερος, γιατί πιέζει ο χρόνος, έχουμε κάπως καθυστερήσει. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, με έχουν καλύψει οι προλαλήσαντες, δεν έχω να πω σπουδαία νέα πράγματα. Υποστηρίζω πάντως τους συναδέλφους μου όσον αφορά την εκπροσώπηση των γυναικών. Νομίζω ότι όντως αυτό το οποίο υπόθηκε ήταν ε, πάρα πολύ σημαντικό το να καταφέρουμε δηλαδή να εξασφαλίσουμε ότι σε μελλοντικέ αντιπροσωπείε θα έχουμε συμμετοχή γυναικών. Ενδεχομένω η γραμματεία να μπορούσε να επιθυμήσει στου συντονιστέ κάθε φορά που διορίζουν μέλη για αντιπροσωπείε να προσέχουν επίση και την εκπροσώπηση των δύο φύλων και τη συμμετοχή γυναικών. Πρέπει να γνωρίζετε επίση ότι το έργο τη αντιπροσωπεία αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί τον σημαντικότερο δωρητή είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν εκπροσωπείται στις συνεδριάσεις αυτές ε, και η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο παίρνει πολύ σχετικές σημαντικές πολιτικές αποφάσεις όσον αφορά την χρηματοδότηση της αναπτυξιακής βοήθειας. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω ότι μας υποδέχθηκαν πολύ πιο θετικά αυτή τη φορά εμάς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από ό,τι στο παρελθόν τόσο στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από, τη, από τα ίδια τα Ηνωμένα Έθνη. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό από μόνο το αποτελεί σημαντικότατη πρόοδο Σαφώς εμείς θα πρέπει να συμμετέχουμε επικοδομητικά, αυτό ακριβώς κάναμε, αλλά αποκομίσαμε και πολύ σημαντικά διδάγματα. Μάθαμε πολύ περισσότερα πολύτιμα πράγματα από ό,τι θα μαθαίναμε αν μέναμε εδώ πέρα στις Βρυξέλλες. Η όλη εμπειρία λοιπόν ήταν πολύ θετική. Σας ευχαριστούμε κύριε Μίτσελ, σας δίνω το λόγο για να ολοκληρώσετε. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε, καταρχάς να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που πήραν το λόγο κάτι το οποίο δεν είπα στην αρχική μου εισήγηση. Συμφωνώ με όλους ε, όσους συνεχάρισαν την γραμματεία. Πραγματικά η γραμματεία διοργάνωσε πάρα πολύ καλά την επίσκεψή μας, τις επαφές που είχαμε με υψηλόβαθμους αξιωματούχους, με τον πρόεδρο της Παγκόσμιας Τράπεζας για παράδειγμα. Πρέπει να ευχαριστήσω επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης που πραγματικά μας στήριξαν, μας συνόδευσαν και μας βοήθησαν πολύ κατά την παρουσία μας στην ε, Νέα Υόρκη. Θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο βελτιωμένη η συνεργασία μας από ό,τι στο παρελθόν. Το εκτιμούμε ιδιαίτερω λοιπόν αυτό και θεωρώ ότι ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε στο δρόμο αυτό. Και όντω συναντήσαμε δύο φορέ για τον αρμόδιο επίτροπο. Πρέπει λοιπόν να επιμείνω στα σημεία αυτά. Πολύ συχνά είμαστε επικριτικοί σε επαφέ που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οφείλουμε λοιπόν να τονίσουμε και την θετική διάσταση τη συνεργασία μα όταν αυτή ε, υλοποιείται. Νομίζω ότι συντοπίσαμε όλοι ότι ήταν ιδιαίτερα επικοδομητική επίσκεψή μας στην Νέα Υόρκη. Πολλοί είχαμε συμμετάσχει στην ενδιάμεση αναθεώρηση της έκθεσης αυτής, αλλά είδαμε ότι να πάμε επί τόπου ήταν πάρα πολύ σημαντικό και πολύτιμο. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή σας, για τον ενθουσιασμό που καταδείξατε, για τις πληροφορίες που μας δώσατε για τους αναπτυξιακούς στόχους χιλιετίας. Έχετε όλοι απόλυτο δίκιο. Θα ήθελα απλώ να κάνω την εξή διευκρίνηση. Εγώ δεν μπόρεσα να συμμετάσχω στην αντιπροσωπή αυτή. Ήμουνα την περίοδο εκείνη στο Αφγανιστάν και ήμουνα επικεφαλής της Επιτροπής Παρακολούθησης των Εκλογών στο Νεπάλ. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι η χώρα αυτή που είναι μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου Όσον αφορά την καταγραφή των ψήφων, προβλέπεται ότι μπορεί να καταγραφεί κανείς στους εκλογικού καταλόγους ως άνδρας, γυναίκα ή προβλέπεται ακόμα και δυνατότητα του δέτερου τρίτου γένους. Θεωρώ λοιπόν ότι ε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό πραγματικό επίτευγμα γιατί υπάρχει πραγματικά μια, ένα ποσοστό του πληθυσμού το οποίο κατεγράφει στους εκλογικού καταλόγους χρησιμοποιώντας τη νέα αυτή δυνατότητα που δίδεται στη χώρα αυτή και το λέω αυτό στον κύριο Γκούσταυσον και στους άλλους οι οποίοι αναφέρθηκαν στην εκπροσώπηση των φίλων. Να δώσω τώρα, τώρα το λόγο στην εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Πάρμπαρα Λούτεν. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ επίσης για τα θετικά σχόλια που κάνατε, για την επίσκεψή σας και για την διοργάνωση την οποία επεφύλαξε για σας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα διαβιβάσω τα θετικά σας σχόλια στους συναδέλφους μου πολύ σύντομα να αναφερθώ στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διάσκεψη αυτή στη Νέα Υόρκη. Χαιρόμαστε και εμείς πάρα πολύ για τη δυνατότητα αγόρευσης που δόθηκε τόσο στον κύριο Πίλμπαξ όσο και στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μπαρόζο, αλλά επίσης και στους άλλους επιτρόπους οι οποίοι μπόρεσαν να πάρουν το λόγο και να τοποθετηθούν κατά τη διάρκεια της υψηλόβαθμης αυτής διάσκεψης στη Νέα Υόρκη. Αυτό ήταν πάρα πολύ θετικό. Πήραμε το λόγο πολύ γρήγορα κατά την έναρξη της συνεδρίασης αυτής και όχι σε διαφορετικά πάνελ και πολύ αργά κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Αναφερθήκατε σε κάποιες πολύ θετικέ εξελίξεις, καθώς επίσης και σε κάποια πολύ θετικά σημεία της έκθεσης αυτής. Το κείμενο αποτελεί, θεωρούμε, μια πολύ θετική εφετηρία στις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις που μας περιμένουν τους επόμενους μήνες και τα επόμενα χρόνια Συμφωνούμε μαζί σας ότι ένα πολύτιμο στοιχείο της έκβασης αυτής είναι η απόφαση που ελήφθη ότι η αναθεώρηση των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας θα λάβει χώρα σε συνδυασμό με τα συμπεράσματα του Ρίο συν 20 και ότι θα πρέπει να συγχωνευτούν, να συγκεραστούν οι στόχοι και τα επιμέρους συμπεράσματα. Επομένως, εκ του σύνεγγυς θα παρακολουθήσουμε εμείς τη διαδικασία για να εξασφαλίσουμε κάτι τέτοιο, όπως είπε ο πρόεδρος Μπαρόσο στην επιστολή του προς τον πρόεδρο Σούλτ στις 11 Σεπτεμβρίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να συνεχίσει να διαμορφώνει την ατζέντα για μια φιλόδοξη συνέχεια όσον αφορά τους αναπτυξιακούς στόχους χιλιετίας χιλιετίας και θα πρέπει αυτό να συνδυαστεί με τους νέους αναπτυξιακούς στόχους χιλιετίας, τους ε, SDGs. Ξέρετε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ρητός έχει αναφέρει στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2014, το οποίο εγκρίθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, στις 22 δηλαδή Οκτωβρίου, ότι προτίθεται να εγκρίνει ένα νέο σύστημα ενημέρωσης και επικοινωνίας κατά το πρώτο εξάμεινο του 2014 όσον αφορά την απτυξιακή βοήθεια. Δεν έχουμε ένα σαφές ακόμα χρονοδιάγραμμα γιατί αυτό θα εξαρτηθεί από τις διεθνείς προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις που θα λάβουν χώρα. Ω προ την ουσία τώρα, στην επόμενη ανακοίνωση Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να πετύχουμε την κατάλληλη ισορροπία ανάμεσα στην υποβολή κάποιων ιδεών που θα τροφοδοτήσουν την όλη συζήτηση και σε ένα υψηλό επίπεδο ευελιξία και διαλλακτικότητα που θα πρέπει να καταδείξουμε ω προ του άλλου συμμετέχοντε στη συζήτηση αυτή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να είμαστε σε θέση να ακούμε και να αφουγκραζόμαστε και του εταίρου μα. Επ' αυτού θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε τις, στις 27 και 28 Νοεμβρίου τις ημερίδες αναπτυξιακής συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίζω ότι θα συμμετέχετε σε αυτές και θα έχουμε μια καταπληκτική ευκαιρία κατά τη διάρκεια των ημερίδων αυτών να ανταλλάξουμε απόψεις με πολλά εμπλεκόμενα μέρη. Περιμένουμε περίπου 50.000 συμμετέχοντες από όλες τις πλευρές του κόσμου και θα συνεχίσουμε και τη συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει με τα ίδια τα κράτη-μέλη τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να καταφέρουμε να εμβαθύνουμε την προσέγγισή μας σε κάποια βασικά στοιχεία για το θεματολόγιο μετά το 2015, για την εξέλιξη δηλαδή των στόχων μετά το 2015. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας με κάποιες σημαντικές χώρες, χώρες κλειδιά. Αυτό έχουμε κάνει στο παρελθόν και αυτό προβλέπεται και για το μέλλον. Αυτά είχα να σας πω. Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να καταβάλω κάποιες θετικές εντυπώσεις σε σχέση με αυτά τα οποία είπαν οι προλαλήσαντες. Σας ευχαριστούμε κυρία Μπάρμπαρα Ντούκε. Το λόγο έχει τώρα λόγος ο κύριος Τζοβάνι Μαστροτσάκομο. Ευχαριστώ πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Σε ζητώ συγγνώμη, αλλά μόλις ανέλαβα την Προεδρία, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάπως ε, παράξενη για μένα αυτή η κατάσταση. Πάντως, αν θέλετε, ευχαρίστως να σας ακούσουμε. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και διαδικασίες που υποστηρίζουν τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την πρόσβαση των αγαθών και υπηρεσιών της Ένωσης στις αγορές δημοσίων συμβάσεων τρίτων χωρών. Μόλις μου είπαν ότι η κυρία Σαρζιχεντίνη που είναι η συγγήτρια ζήτησε να προσθέσουμε και άλλο ένα σημείο, δηλαδή τη συζήτηση περί των για την οδηγία της όσον αφορά την αποκάλυψη μη οικονομικών πληροφοριών. Σχέδιο χνομοδότησης που πρέπει να ψηφιστεί σήμερα το απόγευμα. Άρα λοιπόν μου ζητάτε να γίνει η συζήτηση των δύο σημείων ταυτόχρονα. Εάν συμφωνείτε βέβαια θα προχωρήσουμε έτσι. Ωραία λοιπόν, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση, καλό την κυρία Σαρσεντίνη να μας πει, να μας κάνει την εισήγησή της. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι και τα δυο μπορούν να είναι πολύ σύντομα. Να κάνω πρώτα το ένα να περιμένω τις απαντήσεις και μετά να περάσω στο δεύτερο. Αν συμφωνείτε. Να ξεκινήσουμε με την πρόσβαση των, ε, τρίτων, ε, των ε, αγαθών και υπηρεσιών τρίτων χωρών στην εσωτερική αγορά της Ένωσης και σχετικές διαδικασίες. Ίσως θα θυμάστε πως η πρότασή μου για γνωμοδότηση της ΔΕΔΕ προς την Επιτροπή ΙΝΤΑ ναι, ήταν να ε, με στόχο να προτείνουμε στην Επιτροπή ήταν να παραπέμψει αυτή την πρόταση πίσω στην Επιτροπή. Και αυτό γιατί δεν πιστεύω πως ο τρόπος με τον οποίο διατυπώνεται η πρόταση της Κομισιόν θα ωφελήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες. Αντίθετα, εξακολουθούμε να βλέπουμε πως οι δημόσιες προμήθειες στον ΠΟΕ δεν ε, εξετάζονται ως ένα φυσιολογικό θέμα εμπορίου και δεν υπάρχουν αναπτυσσόμενε χώρε που το συνυπογράφουν. Την περασμένη σύνοδο, μία μόνο αναπτυσσόμενη χώρα υπέγραψε σε αυτή τη σύμβαση, που ήταν η Αρμενία. Αλλά θα σα θυμίσω πω είναι διαφορετική περίπτωση, γιατί η Αρμενία προσπαθεί να βρει τη θέση της ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την πρώην Σοβιετική Ένωση. Η πρόταση για τις δημόσιες προμήθειες και την αμοιβαιότητα έχει στόχο τις χώρες BRICS, αλλά στην πρότασή της η Κομισιόν ασχολείται με όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες που δεν είναι λιγότερο αναπτυγμένες χώρες, LDC. Είχα μια συζήτηση με τον Επίτροπο Μπαρνιέ ε, για θέματα εσωτερικής αγοράς, ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε και να το αλλάξουμε αυτό. Εγώ εκτίμησα αυτή τη, τα λόγια, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει αλλάξει κάτι. Κατά τη γνώμη μου, η πρόταση ως έχει δεν θα έχει κανένα πρακτικό αποτέλεσμα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως προστασία των δικών μας αγορών, αλλά και για να αναγκάσει να ανοίξουν αγορές αναπτυσσόμενους χωρών, ενώ θεωρώ πως οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίζουν αν θα χρησιμοποιούν τις δημόσιες προμήθειες ως κίνητρο, ως βοήθεια για τις τοπικές αγορές. Τούτου λεχθέντος, οι περισσότερες τροπολογίες που υποβάλλατε με βρίσκουν σύμφωνοι, αλλά τελικά θα, τις καταψη... θα καταψηφίσω ούτως ή άλλως την πρόταση. Εάν δεν με ακολουθήσετε, που είναι δικαίωμά σας, θα πρέπει να γνωρίζετε απλά πως εγώ ως εισηγήτρια δεν θα υποστηρίξω την πρόταση αυτή στην γνωμοδότηση προς την Αυτή είναι η πρώτη έκθεση, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κάποιος να πάρει το λόγο. Όχι. Σιωπάτε. Ε, και εγώ θέλω να θέσω μια ερώτηση στην Κομισιόν, αφού ακούσαμε την κυρία Σταρζεντίνη που μας ε, ε, ενημέρωσε για τους φόβους της όσον αφορά την εξέλιξη αυτού του φακέλου. Μπορώ να συναψίσω τη θέση σας με, ως εξής, ότι δηλαδή θα μπορούσε να γίνει μια παράκαμψη σε σχέση με την ε, βοήθεια που προορίζεται σε συγκεκριμένα κράτη. Ε, θα δώσω το λόγο στην Κομισιόν και στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για να απαντήσει στα ερωτήματά μας και, και στα ερωτήματα της κυρίας Αρζεντίνη. Ε, κύριε Πρόεδρε, εγώ προέρχομαι από την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Καταρχήν ένα γενικό σχόλιο για την πρόταση της Κομισιόν. Θεωρείτε πως είναι πολύ σημαντικό να ανοίξουν οι ε, ξένες ε, αγορές δημοσίων συμβάσεων και είναι ένα από τα πιο σημαντικά θέματα όσον αφορά τις συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου για να προωθήσουμε δηλαδή το μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων. Αυτό δεν είναι πολύ εύκολο και η Κομισιόν πιστεύει πως ένα εργαλείο μόχλευσης είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και έχουμε υποβάλει αυτή τη σημαντική πρόταση. Θα ήθελα να υπογραμμίσω εντόνως ότι δεν είναι άποψη της Κομισιόν ότι θα πρέπει να στοχεύουμε τις στοχότερες χώρες. Αντίθετα, οι μεγαλύτεροι εμπορικοί εταίροι είναι αυτοί που έχουν ε, κάνει διακρίσεις κατά των ευρωπαϊκών εταιριών και για αυτούς προσπαθούμε να ασκήσουμε πίεση. Να έχουμε δηλαδή θέλουμε ένα εργαλείο όχι προστατευτικό, θα πρέπει να ανοίξουν η αγορά σημαντικών μεγάλων τρίτων χωρών, πλούσιων τρίτων χωρών που διαρκώς κάνουν διακρίσεις εναντί των Ευρωπαίων ε, ε, επιχειρηματιών. Θα, βέβαια θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι μικρότερες, ε, μικρότεροι φορείς, οι μικρομεσαίες της αναπτυσσόμενης χώρας δεν θα πληθυγούν από αυτήν εδώ την πρόβλεψη. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να δούμε τη διαδικασία που θα είναι μία έρευνα πολύ προσεκτική ώστε να ελέγξουμε αν υπάρχουν ή όχι διακρίσεις και επίσης θα υπάρχει διαδικασία διαβούλευσης προηγουμένως και φυσικά η ιδέα διαβουλησης προηγουμενως και φυσικα η ιδεα ειναι πως το μέτρο αυτό θα πρέπει να θεσπιστεί και φυσικά ε, θα πρέπει να γίνει σημαντικός διάλογος και διαπραγματεύσεις. Έγιναν αναφορές τώρα στην ενίσχυση και στην αναπτυξιακή βοήθεια, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε πως αυτά τα κονδυλία δεν έχουν καλυφθεί από τις οδηγίες της Κομισιόν και ούτε από αυτό εδώ το μέσο. Δεν είναι στόχος του μέσου να προτείνει ότι η ε, αναπτυξιακή βοήθεια δεν θα πρέπει να σέβεται τις ευρωπαϊκές δεσμεύσεις όσον αφορά την αποτελεσματικότητα. Αντίθετα, το μέσο αυτό τονίζει τη σημασία της καταπολέμησης των διεφθαρμένων πρακτικών μέσω ενός διαφανούς προγράμματος δημοσίων συμβάσεων. Δίνω το λόγο στον συνάδελφό μου για να συμπληρώσει. Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον πρόεδρο που μας έδωσε το λόγο. Θα ήθελα και εγώ να τονίσω πως δεν είναι πρόθεση της Κομισιόν και της προτασής της να οδηγήσει σε περιορισμό της ενίσχυσης γιατί βεβαίως... Δεν είναι πρόθεσή μας να δώσουμε αυτή τη βοήθεια υπόρους και προποθέσει ένα στενότερο πλαίσιο και σε αυτό το πλαίσιο μπορώ να πω ότι αυτή η πρόταση δεν θα ίσχυε για την αναπτυξιακή βοήθεια από την ε, Γενική Διεύθυνση ΑΦΚΟ και για την ε, επίσημη βοήθειά μας ε, και αυτό δεν θα οδηγούσε σε αύξηση περιοριστικών πλαισίων. Το ίδιο ισχύει για το ότι δεν θέλουμε να υπάρξει οποιαδήποτε επίπτωση όσον αφορά τις τη διαφοροποίηση αναπτυσσόμενων χωρών όταν θα έχουμε ε, με την ανάθεση έργου, εκτέλεση έργου. Θα, είναι, ε, θα έχουν τη διακριτική ευχαίρεια να χρησιμοποιούν και τις δικές δυνατότητες. Επίσης, να τονίσω στο τέλος ότι αυτή η πρόταση δεν στοχεύει στο να στοχοθετήσει, στοχοποιήσει αναπτυσσόμενες χώρες ε, και μπορώ να επαναλάβω μόνο αυτό το οποίο ανέφερε ήδη στο παρελθόν ο Επίτροπος Μπανέ, ότι είναι ανοιχτή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε προτάσεις που μπορούν να βελτιώσουν τα μέσα και τα εργαλεία σε σχέση με αυτές τις δυνατότητες. Σημειώνουμε κάποιες τροποποίησεις και τροπολογίες που έχουν κατατεθεί από τη δική σας Κοινοβουλευτική Επιτροπή που θα επέκτηνε την, τον κατάλογο των αποκλειόμενων χωρών, πράγμα το οποίο φυσικά θα αύξαινε σημαντικά το εύρος ε, όσον αφορά τις ε, ε, μη αποδεκτές χώρες, αναπτυσσόμενες χώρες και αναγνωρίζουμε φυσικά μέσα σε αυτό το πλαίσιο ότι αυτή η πρόταση έχει την χάρη της υποστήριξης και άλλων κοινοβουλευτικών επιτροπών επίσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε που απαντήσετε στα όσα είπε η κυρία Σαρτζεντίνη. Ο κύριος Γκούσταυσον έχει τώρα το λόγο. Πρωτού δώσω το λόγο πάλι στην κυρία Σαρτζεντίνη. Ο κύριος ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο Σαρτζεντίνη όσον αφορά το, την τελική αυτή έκβαση του εγγράφου. Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να καταλάβω πάρα πολύ καλά το ζήτημα. Βλέπω ότι η πρόταση έχει να κάνει με την ανάπτυξη, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να υποστηρίξουμε το επιχείρημα αυτό το οποίο έχουμε στην έκθεση αυτή, ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται τελικά είναι δικαιολογημένα, εφόσον δεν προτείνονται από την ενδιαφερόμενη τελικά χώρα. Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στις διάφορες συναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά την πρόσβαση στις δημόσιες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να εξαναγκάσουμε τις χώρες ε, και για την ε, εξίσωση, ισότητα μεταξύ δυτικών και ανατολικών χωρών. Δηλαδή τι θα κάνουμε, θα επιβάλλουμε υποχρεωτικά σε αυτές τις χώρες κάτι. Όπως η ίδια κυρία Σαρτζεντίνη προανέφερε, εμείς οι ίδιοι αυτά τα θέματα σε σχέση με τις δημόσιες ε, ε, προσφορές και ε, συμβάσεις έχουμε απορρίψει ένα τέτοιο πλαίσιο και μπορεί κανείς να σκεφτεί οτιδήποτε ακόμα και αν σκέπτεται κανείς ότι μια τέτοια ρύθμιση είναι καλή πώς μπορεί να πει στους άλλους αν εμείς θεωρούμε κάτι ότι δεν είναι καλό και δεν θεωρείται προς όφελός τους πώς μπορούμε να τους το επιβάλλουμε ας φανταστούμε ότι μπορεί να, βρισκόμαστε, να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση σε σχέση με την ανάπτυξη των χωρών της Δύσης σε κοινωνικά κράτη ευημερία ευημερίας και πρόνοιας. Αν κάτι μας επιβαλόταν εκ των έξω τότε τι θα κάναμε, δεν θα είχαμε αναπτυχθεί ποτέ με αυτόν τον τρόπο. Και αν λέει κανείς ότι τώρα οι αγορές πρέπει στις αναπτυσσόμενες χώρες να ανοίξουν και να λειτουργούν όπως στις δικές μας χώρες, αυτό μπορεί να γίνεται μόνο αν είμαστε ισότιμοι ή ίσοι εταίροι. Δεν είμαστε όμως ισότιμοι και ίσοι εταίροι. Ελπίζω δεν θα υπερψηφιστεί αυτό το σημείο. Ευχαριστώ. Κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Άκουσα προσεκτικά αυτά τα οποία ανέφερε στην παρέμβασή της αυτή τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε προηγούμενες, ε, με προηγούμενες ευκαιρίες. Ε, αυτή η πρόταση δεν έχει καλά διατύπωθεί και δεν έχουμε προβληματιστεί επαρκώς ποιες επιπτώσεις θα υπάρξουν στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ε, πιστεύω επίσης ότι αυτή, αυτή η πρόταση τη συζήτηση στον ΠΟΕ, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, τη συζήτηση για τα θέματα των δημόσιων συμβάσεων την υπονομεύει δεν γίνεται χωρίς λόγο για το ότι δηλαδή δεν θα αποτελούν ε, μέρος των διαπραγματεύσεων ε, οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες και αυτό δεν είναι καλό και το πώς θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε ένα θέμα αποτελεσματικότητας στις δράσεις. Πάλι τίθεται το θέμα για τις αγορές προμηθειών και τις συμβάσεις προμηθειών. Για το ότι εδώ θα έχουμε όρους ή προϋποθέσεις που θα ισχύουν για την αναπτυξιακή βοήθεια. Πρέπει να πω ειλικρινά και ανοιχτά. Σε αυτή τη χρονική στιγμή όταν είχαμε σε συζήτηση διμερή και μας είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν από δύο εβδομάδες ότι αυτό κάπως πλημελώς έχει διατυπωθεί και πρέπει να διαφοροποιηθεί και όταν λέμε από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τώρα ότι οι αναπτυσσόμενες ε, χώρες ε, ε, και οι λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες θα είναι θύμα αυτής της κατάστασης τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να το προσέξει και να ανταποκριθεί. Σας ευχαριστώ κυρία Σαρτζεντίνη. Τώρα μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις τροπολογίες σας όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης για την οδηγία κοινοποίησης των μη οικονομικών πληροφοριών των εταιριών, ε, έκθεση την οποία θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η γνωμοδότηση την οποία συντάσσουμε ουσιαστικά εντάσσεται στη γενικότερη συζήτηση την οποία διεξάγουμε για την διαφάνεια των πολυεθνικών εταιριών που ουσιαστικά έρχεται σε συνέχεια με την, από την ψηφορία που είχαμε για την οδηγία για την διαφάνεια των εταιριών αυτών. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ θετικό το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αποφασίσει να νομοθετήσει για την κοινοποίηση των μη οικονομικών πληροφοριών των εταιριών αυτών και είμαι υπέρ των τροπολογιών που έχουν υποβάλει οι συνάδελφοί μου, κυρίως από την ΑΛΔΕ, όπου ενισχύουν και διευκρινίζουν όλη τη διατύπωση που χρησιμοποιείται για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς επίσης και όλες τις πληροφορίες που τις μη οικονομικές πρέπει να παρέχονται από τις εταιρείες. Επίσης, οι σοσιαλδημοκράτες προσπαθούν ε, να ενισχύσουν κάπως τη διατύπωση όσον αφορά τα μέτρα κατά της διακρατικής μεταχείρισης και έχουμε και προτάσεις από το ΕΛΚ πάλι για την εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς επίσης και για τις κοινωνικές επενδύσεις και τα κοινωνικά κριτήρια. Θεωρώ πραγματικά ότι οι προτάσεις σας, αγαπητοί συνάδελφοι, καθιστούν τη γνωμοδότησή μας πολύ πιο ισχυρή. Υπάρχουν ε, βέβαια δύο συμβαστικές λύσεις τις οποίες έχω καταλήξει, δύο συμβαστικές τροπολογίες, όπου από ό,τι βλέπω δεν μπορούν να συμφωνήσουν οι συνάδελφοι από το ΕΛΚΑ. Πρώτον, ο ορισμός για το τι είναι μικρομεσαία επιχειρήση. Άλλαξα τη σχετική διατύπωση στην πρόταση και ουσιαστικά έχω κάνει λιγότερο περιοριστική την, τον ορισμό αυτό, ώστε να συνάδει με την οδηγία για τα λογιστικά πρότυπα τα οποία, ε, την οποία εγκρίναμε τον προηγούμενο Ιούνιο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα σας βρει ο νέος αυτός ορισμός και γενικότερα προτάσεις μου σύμφωνους. Εν γέννη θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους ιδιαίτερως για την υποστήριξή σας, για τη βοήθειά σας και για το ότι με τη συμβολή σας κάνετε τελικά πολύ πιο στεναρή τη γνωμοδότηση αυτή. Προσβλέπω λοιπόν στη δική σας υποστήριξη. Σας ευχαριστώ και πάλι. Eh σας ευχαριστούμε κυρία Σαρτζεντίνη. Υπάρχουν μέλη της Επιτροπής μας που θα θέλουν να πάρουν το λόγο. Γκέι Μίτσελ. Κύριε Πρόεδρε, σε σχέση με τον ορισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πρωτού ψηφίσουμε το απόγευμα, Πρόεδρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να πάρει το λόγο δεν παρίσταται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν έχει εκπρόσωπο το σημείο αυτό, καθότι ε, προσθέθηκε τελευταία στιγμή. Σα ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο τη μερίσιας διάταξη, το επαριθμόν 12, έκθεση τη κυρία Κρετού. Ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης της κυρίας Κρετού προς την Επιτροπή των Γυναικών για την σεξουαλική εκμετάλλευση και εκπόρνευση και τις επιπτώσεις του στην ισότητα των φύλων. Κυρία Κρετού, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε το σχέδιο γνωμοδότησή σας. Σα ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Χαρά μου είναι να παρουσιάσω λοιπόν τη γνωμοδότηση αυτή που συντάχθηκε από την δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και την Ισότητα των Φίλων. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό η σεξουαλική εκμετάλλευση, η πορνεία και η βία. Είναι πολύ σημαντικά προβλήματα και οι καταχρήσεις ε, εδώ σημαντικών θεμελιωδών δικαιωμάτων και σε σχέση και με την οικονομική και την ε, περιφερειακή και κοινωνική κατάσταση των θυμάτων. Τα θύματα αυτής της βίας είναι συνήθως κορίτσια, γυναίκες και παιδιά που δεν έχουν το κοινωνικό και οικονομικό καθεστώς να αντισταθούν ή να αποφύγουν αυτή την κατάσταση. Ιδιαίτερα τα νερά κορίτσια για αυτές τις καταχρήσεις ε, όσον αφορά και την οικιακή οικογενειακή βία, την, ε, <clears throat> τον, τους βιασμούς, ε, την σεξουαλική εκμετάλλευση, τον ακροτεριασμό γεννητικών οργάνων και η, ανθρωπο, η ανθρωποεμπορία, η εμπορία ανθρώπων είναι και αυτή είναι ένα φαινόμενο που συνδέεται γενικότερα με αυτά και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι θεσμοί της, οι εθνικές κυβερνήσεις και όλοι οι οργανισμοί και οι εμπλεκόμενοι πρέπει να συνεργαστούν για την δημιουργία κοινών όρων και προϋποθέσεων για την εγκληματοποίηση, την καταδίωξη και την ε, ποινική κύρωση αυτών των αδικημάτων ε, και σε σχέση και με τις διακριτική, τη διακριτική μεταχείριση που έχει επιδεινωθεί και οδηγεί σε αυτές ε, τις σημαντικές παραβιάσεις που οδηγούν σε σημαντικά τραύματα σωματικά και ψυχικά για τα θύματα. Έχουμε κάποιες προτάσεις που υποβάλλουμε προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας Φύλων να συμπεριληφθεί το, στην πρόταση ψηφίσματος ε, να συμπεριληφθούν κάποια θέματα. Πρώτα απ' όλα ζητούμε οι κυβερνήσεις να μειώσουν το κόστος ε, για την υγεία και τους ελέγχους και τις εξετάσεις ε, ε, και έχουμε ζητήσει να βοηθηθούν τα θύματα, τα κορίτσια, τα παιδιά, οι γυναίκες που ανήκουν σε μειονότητες ιδιαίτερα να βοηθηθούν. Η διαφθορά είναι επίση ένα θέμα, για τον λόγο αυτό συνεχίζει να υπάρχει η εμπορία ανθρώπων και παραμένουν ατιμόρυτοι υπεύθυνοι. Η διαφθορά εδώ διαδραματίζει ένα ρόλο όσον αφορά την εμπορία και αυτά τα φαινόμενα. Θέλουμε να υπάρξει Κράτο κράτος δικαίου και σωστή διαχείριση και διακυβέρνηση στα κράτη, τα ε, αδικήματα αυτά πρέπει από κοινού να διώκονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη για να αντιμετωπιστούν όπως πρέπει. Ανάπτυξη υπηρεσιών στις αναπτυσσόμενες χώρες, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων, είναι ένα άλλο πρόβλημα, το οποίο έχει επιπτώσει σε αυτά τα, σε αυτά τα άτομα. Η σεξουαλική εκμετάλλευση θα πρέπει να αποτελεί αντικείμενο αποτελεσματικών κυρώσεων και διώξεων, αποτελεσματικών ποινών χωρών αποτρεπτικών ποινών και πρέπει τα θύματα να τα επικουρούμε για όσο χρονικό διάστημα είναι αναγκαίο να γίνεται αυτό για τη σωματική τους και ψυχολογική τους ανάκτηση και αποκατάσταση. Πρέπει να βρούμε τις πιο ενδεδειγμένες λύσεις για να αντιμετωπιστούν όλες οι μορφές βίας και διακριτικής μεταχείρισης εις βάρος των γυναικών, των κοριτσιών και των παιδιών και όλες οι μορφές βίας ε, να καταργηθούν και να καταπολεμηθούν ιδιαίτερα για τα πιο ευαίσθητα ε, θύματα που είναι γυναίκες και αντιμετωπίζουν αυτά τα προβλήματα. Ευχαριστώ για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Κρετού. Θα δώσουμε το λόγο στην κύριο Γκούσταυσεν και μετά στην κύριο Γκέι Μίτσελ. Σας ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ την κυρία Κρετού για μια πάρα πολύ καλή γνωμοδότηση και πραγματικά ευελπιστώ και μπορώ να πω ότι η έκθεση αυτή στην Επιτροπή ε, Δικαιωμάτων των Γυναικών θα μπορέσει να βελτιώσει τα πράγματα και να ληφθεί υπόψη. Δεν έχω καμιά αντίρρηση ή ένσταση έναντι αυτών που προανέφερε η συνάδελφος. Έχω όμως κάποια πράγματα που θα ήθελα να προσθέσω και όσον αφορά και τροπολογίες σε σχέση με αυτά τα οποία αναφέρατε και θα πρέπει να ενδυναμωθούν κάποια θέματα για την πρώτη παράγραφο, παράγραφο 1. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό η διασύνδεση μεταξύ πορνείας και εμπορίας ανθρώπων να καταστεί να διαφρύνει διευκρινιστεί. Αν δεν υπήρχε ζήτηση από πλευρά των ανδρών, δεν θα υπήρχε πώληση τέτοιων υπηρεσιών και δεν θα υπήρχε το φαινόμενο της πορνείας. Επίσης ε, έχουμε έχω μια τροπολογία που θέλει να αποσαφηνίσει ότι τα κύρια αίτια έγινε στο ότι έχουμε έναν άνισο κόσμο, ένα κόσμο με πολύ μεγάλες ανισότητες, ε, με ματριαρχικές δομές, ε, σε κάποιες περιπτώσεις ή πατριαρχικές σε άλλες και πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Επιπλέον, αυτό το οποίο ήδη αναφέρατε και πρέπει να ενδυναμωθεί περαιτέρω είναι το ότι οι ε, πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σε μειονεκτική θέση, ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες και ε, μειονότητες πρέπει να υποστηριχθούν με κάθε τρόπο. Και αυτό αφορά και την επιλογή των όρων και της ορολογίας. Πρέπει να κάνουμε ρόλο για αρνητική διακριτική μεταχείριση. Δεν είναι ευάλωτα, ευάλωτες οι γυναίκες μόνο, βρίσκονται και σε μειονεκτικές θέσεις. Δεν είναι η θέση τους μόνο, αλλά έχουμε disadvantage που πρέπει να χρησιμοποιείται μειονεκτική θέση ε, αντί vulnerable, αντί εύθρωτοι, ευάλωτοι. Και επίσης ε, για τις γυναίκες πρέπει να ισχύουν σε ε, περιοχές συγκρούσεων και σειράξεων ε, δυνατότητες που θα λαμβάνουν υπόψη αυτή την κατάσταση και θα τις βοηθούν. Στην παράγραφο 3, παράγραφο 3 στη συνέχεια, εδώ γίνεται λόγος για σεξουαλική βία. Είναι σημαντικό αυτό όμως από την άλλη πλευρά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι τέτοιου είδους ε, βία χαρακτηρίζει πολλές φορές ε, τις σχέσεις μεταξύ γυναικών ανδρών ε, αλλά και αντίστροφα στην κοινωνία μας. Όμως το μεγαλύτερο τμήμα αυτής της βίας προέρχεται από τους άνδρες κατά των γυναικών. Γι' αυτό λέω mostly by men against women. Δηλαδή τις περισσότερες φορές από τους άνδρες εις βάρος των γυναικών. Και έχει δίκιο η, η συντάκτρια γνωμοδότηση χρηματοδότησης ότι χρειάζονται εθνικά προγράμματα και σχέδια για να σημειωθεί πρόοδος. Σε αυτά τα ε, προγράμματα και σχέδια ε, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τον σεξουαλικό τουρισμό για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Αν δεν υπήρχε ζήτηση δεν θα υπήρχε και αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ. Uh, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ για αυτή την έκθεση και τη μάλλον γνωμοδότηση που υποστηρίζουμε βεραίως. Και θα δούμε και τις τροπολογίες μετά από την, το πέρας της προθεσμίας. Νομίζω πως είναι σημαντικό το θέμα και πως η γνωμοδότηση ε, ε, ε, αντιμετωπίζει τις ανησυχίε που έχουμε για το θέμα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει τώρα ο κύριος Ρικάρτο. Είναι εκπρόσωπος της ε, Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Ε, πιστεύουμε πως ε, συμφωνεί με τις γραμμές της πολιτικής μας όσον αφορά την καταδίκη κάθε είδους βίας κατά των γυναικών καθώς και την παρεμπόδιση της πλήρους άσκησης των δικαιωμάτων τους. Έχουμε κάνει συντονισμένες προσπάθειες Προσπαθούμε κάθε φορά να παρεμποδίσουμε την σεξουαλική εκμετάλλευση. Ε, να σας αναφέρω την 57η ε, Σύνοδο της Επιτροπής για την κατάσταση των γυναικών στον ΟΗΕ όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μια βιώσιμη προσέγγιση κατά των, ε, ε της εκμετάλλευσης των γυναικών όσον αφορά τη δική μας πολιτική σε σχέση με τους εταίρους μας να αναφέρω τις κατευθυντήριες γραμμές της Ένωσης για το τέλος της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών καθώς και το στρατηγικό πλαίσιο δράσης για την ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία που υιοθετηθήκε το 2011 είναι πιο πρόσφατο και είναι το γενικό μας, η γενική μας βάση όσον αφορά την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ολόκληρο τον κόσμο. Και έπειτα να σας αναφέρω και τη συνεργασία που ε, έχουμε αναπτύξει με την Κομισιόν και να δώσω το λόγο στο συνάδελφο από την ε, DG Home που γνωρίζει περισσότερα ε, για τα όσα κάνουμε στον τομέα της ελευθερίας της δικαιοσύνης και της ασφάλειας και δικαιοσύνης. Εγώ γενικά να πω πως συνεργαζόμαστε με τις υπηρεσίες της Κομισιόν για να εξασφαλίσουμε τα, ότι λαμβάνονται υπόψη τα γυναικεία δικαιώματα σε όλες τις υποεπιτροπές για την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη στις οποίες εργόμαστε σε επαφή με τρίτες χώρες. Και τώρα θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο από την ε, Γενική Δεύση ΧΟΜ. Είναι η κυρία Φρεντερίκ Φραστρέ, όχι. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Με συγκεκριμένη επικέντρωση στην εμπορία ανθρώπων και την εξωτερική διάσταση αυτής της ανθρωποεμπορίας και ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα ανάπτυξης. Θα ήθελα να τονίσω με έμφαση ότι η πρόσφατα εγκριθήσα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκρίζωση της ανθρωποεμπορίας ταυτοποιεί ως αίτια, ως ρίζες αυτού του εμπορίου την ανισότητα μεταξύ των φύλων, διακριτική μεταχείριση όσον αφορά τις γυναίκες, σειράξεις, συγκρούσεις και ανασφαλές πλαίσιο μέσα στο οποίο ζουν οι γυναίκες. Όσον αφορά την ανθρωπομορία, για να τονίσω κάποια πράγματα, εργάζομαι για το συντονιστικό όργανο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην GD Home για την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου. Ένα μέρος της εντολής είναι ο συντονισμός των πολιτικών μας στην εξωτερική διάσταση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, κατευθυντήρια γραμμή είναι το έγγραφο προσανατολισμών και που η δεύτερη έκθεση εφαρμογή πρόσφατα εγκρίθηκε από το Συμβούλιο και ταυτοποιεί δέκα προτεραιότητες και όσον αφορά και χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες σχεδιάζουμε στενή συνεργασία. Καθώς επίσης και για το συντονιστή τον ίδιο που εμπλέκεται και συνεργάζεται σε σχέση με αυτές τις 10 χώρες προτεραιότητες για να συνεργαστούμε σε βάθος με αυτές με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ένταση. Το θέμα του φύλου έχει θεμελιώδη ε, ε, ισχύ και σημασία στην καταπολέμηση της ανθρωποεμπορίας. Πολλές φορές ε, έχουμε και την πλειοψηφία ακριβώς αυτών των θυμάτων που είναι ακριβώς οι γυναίκες. 80% είναι γυναίκες αυτού του φαινομένου. Η ευρύτερη εκμετάλλευση ε, σε σχέση με αυτό είναι η σεξουαλική εκμετάλλευση. Ενδιαφέρον είναι ότι 96% των θυμάτων αυτής της σεξουαλικής εκμετάλλευσης του εμπορίου είναι ακριβώς κορίτσια και γυναίκες. Και σε αυτή τη φάση θα ήθελα να αποσαφηνίσω κάτι, να πω ότι έχουμε πολύ καλή συνεργασία επίσης και με την ε, Γενική Διεύθυνση για Συνεργασία για την Ανάπτυξη, εφαρμόζοντας μια ολόκληρη σειρά σχεδίων και προγραμμάτων όσον αφορά την διάσταση καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και σημεία κλειδιά της πολιτικής μας που, ε, ε, συμπεριλαμβάνουν το φύλλο και τις διακριτικές τη διακριτική μεταχείριση κατά των γυναικών λαμβάνονται υπόψη. Ολοκληρώσατε, η κυρία Κρετού έχει τώρα τον λόγο παρακαλώ. Thank you for... Σας ευχαριστώ. για όλα σας τα σχόλια και σας ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κύριο Γκούσταυσον για το έργο για την Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών. Έχει δίκιο, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση οι γυναίκες. Αυτό αληθεύει. Τις καθιστά και ευάλωτες. Θα ήθελα να τονίσω επίσης ότι το φαινόμενο της σεξουαλικής εκμετάλλευσης φτάνει σε ένα κρίσιμο κατόφλι ως επίπεδο για τις αναψώμενες χώρες. Οικονομικά, κοινωνικά, ιατρικά, υπό όλες αυτές τις πτυχές. Διότι σε αυτές τις περιοχές και περιφέρειες αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις οι γυναίκες στην πρόσβαση ακριβώς για την παιδεία και την εκπαίδευση. Έχουν πολύ χαμηλότερους μισθούς και απολαβές και δεν έχουν με κανένα τρόπο πρόσβαση σε υψηλών προδιαγραφών υγειονομική περίθαλψη. Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε εδώ σε αυτό το επίπεδο και φυσικά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εξευρεθούν λύσεις για τη μείωση αυτής της ακραίας παραβίασης δικαιωμάτων του ανθρώπου. Όπως προαναφέρατε προηγούμενα πρόεδρε, η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για αυτή την γνωμοδότηση είναι αύριο, 12 το μεσημέρι ακριβώς. Και σας ευχαριστώ και πάλι λοιπόν. Merci, vous venez déjà faire. Σας ευχαριστώ μόνοι σας λοιπόν κάντε την ανακοίνωση για την προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών. Σας ευχαριστώ. Πρόκειται για τη 12η Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Ολοκληρώνεται η πρωινή μα συνεδρίαση. Συνεχίζουμε σήμερα το απόγευμα στις 3.30, όχι όμως την αίθουσα αυτή, όχι στην αίθουσα αυτή, γιατί δεν έχουμε συσκευές για ψηφοφορία. Θα γίνει λοιπόν αλλαγή αίθουσας για σήμερα το απόγευμα. Θα συνεδριάσουμε στην αίθουσα 6 v Β001. Θα συνεδριάσουμε το παραλαμβάνω στις 3.30 το απόγευμα στην αίθουσα PHS 6 v 001 Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας στην συνεδρίαση αυτή. Καλή σας όρεξη.